Φτάσαμε στο τέλος ημερήσιας διάταξης για απόψε. Να σας υπενθυμίσω πως η συνεδρίαση θα επαναληφθεί αύριο 3η 23 Οκτωβρίου και θα ξεκινήσει σε μια ώρα ασυνήθιστη 8.30 η ώρα με 10 και 20 ένα σύντομο σημεριανό διάλειμμα και μετά βεβαίως ένα διάλειμμα και το απόγευμα και συνέχεια το βράδυ. Η ημερήσια διάταξη